Ε, ο εισηγητής, ο κύριος Γιάβορ, έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι από τις σημαντικότερες εκθέσεις που συζητούμε ετησίως εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο όχι μόνο διότι αφορά χρήμα πολύ δημόσιο χρήμα. Αλλά επίσης σε περιστάσεις δύσκολες που περνάμε τώρα χρειάζεται να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη των ανθρώπων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό για τα θεσμικά όργανα και για κάθε υπεύθυνο ευρωπαϊκό πολιτικό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι χρησιμοποιούνται σωστά τα χρήματά τους με διαφανή τρόπο και δαπανώνται με τρόπο που ταιριάζει με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Η έκθεση που συζητούμε ΥΟΣ εν γέννη αντικατοπτρίζει την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέτος ήταν καλή και ενδελεχής η έκθεση. Το Κοινοβούλιο ως συνήθως έχει δικά του θέματα θέλει να θίξει και δικές του προτεραιότητες. Η έκθεση που ψηφίσαμε στην ε, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου Προπολογισμού έτυχε μεγάλη υποστήριξη από τις πολιτικές ομάδες, ψηφίστηκε σχεδόν ομόφανα στην Επιτροπή. Βασικά επικεντρωνόμεθα επί δύο επιπέδων όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να προστατεύσουμε το εισόδημα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, του ιδίου πόρου αυτή. Από αυτή την έποψη λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να τονίσουμε ότι η απάτη του ΦΠΑ αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διότι το ΦΠΑ ανήκει στους ιδίους πόρους της Ενώσεως και το κενό του ΦΠΑ ποικίλει όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και μεταξύ κρατών μελών. Οι διαφορές μεταξύ ΦΠΑ έφτασαν τα 168 δις ευρώ το 2013. Καλωσορίζουμε την υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει μια στεναρή οδηγία για το ΦΠΑ. Θέλουμε να συμπεριληφθεί και στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να είναι αποτελεσματική προσέγγιση. Εδώ και δύο μέρες περίπου το Ευρωπαϊκό Ελεκτρικό Συνέδριο δημοσίευσε μια ειδική έκθεση όσον αφορά το ΦΠΑ. Υποστηρίζει την άποψή μα. Δηλαδή το σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ενώση για το ΦΠΑ δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό. Τα στοιχεία των κρατών μελών δεν είναι αξιόπιστα. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών δεν λειτουργεί ορθώς και δεν υπάρχει επαρκή συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών. Και η Όλαφ δεν έχει αρμοδιότητα για να διερευνήσει περιπτώσεις ε, διασυνοριακής απάτη στον το ΦΠΑ. Επίση υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Όσον αφορά το ρυθμό ανάκαμψης, το 2014 ήταν 24%. Ε, το ιστορικό ελάχιστο. Και πρέπει να αλλάξει. Το άλλο επίπεδο Προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι δαπάνε πώ χρησιμοποιούνται οι πόροι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν κοινή ευθύνη για την υλοποίηση περίπου το 80% του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτελέσει του προπολογισμού. Άρα έχει πολλά θέματα να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε μια ορθή οικονομική διαχείριση όταν δαπανώνται τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πρέπει να συνάδει με τη βέλτιστη χρήση κάθε ευρώ δεχθήκαμε μια οδηγία για τις ε, κρατικές προμήθειες και τις διαγωνισμούς, αλλά πρέπει να ελέγξουμε πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Ο δείκτης της διαφθοράς αναφέρεται στην έκθεσή μας. Και έχουμε και την έκθεση ε, κατά πολεμής διαφθοράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένεται στο Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι φέτος η έκθεση αυτή θα συμπεριλαμβάνει το 21ο κεφάλαιο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και θέλουμε καλύτερη προστασία για τους πληροφοριοδότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, διότι αυτοί παρέχουν πληροφορίες, επιτελούν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση διαφθοράς. Πιστεύω ότι μαζί με τους κοιόδης εισηγητές ήταν πολύ καλή συνεργασία. Ετοιμάσαμε μια έκθεση η οποία πιστεύω ότι μπορεί να υποστηριχθεί από εσά. Ευχαριστώ. Η κυρία Γεωργίευα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ελέγχου των προπολογισμών και όλο ιδιαιτέρως τον Μπένεντεκ Γιάβορ, τον συγητή για την ετήσια έκθεση 2014 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μα για την ισχυρότατη δέσμευση που έχει αναλάβει το Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση της απάτης. Συμμεριζόμαστε πλήρως αυτή την δέσμευση και καλωσορίζουμε το περιεχόμενο την ανάλυση της έκθεσης καθώς και τις πολύτιμες συστάσεις σας, στις οποίες φυσικά θα δώσουμε συνέχεια. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποιες από τις συγκεκριμένε συστάσεις και τις στάσεις μας σε σχέση με αυτές. Ως προς την καταγραφή των παρατυπιών, το Κοινοβούλιο ζήτησε και δικαίως να αναβαθμιστεί η συγκρισιμότητα των δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να διαμορφώνουμε μία εικόνα που είναι κατανοητή και μας επιτρέπει να αντλήσουμε και συμπεράσματα. Το 2015 υιοθετήσαμε ένα νέο κανονισμό σε σχέση με την υποβολή αναφορών για τις παρατυπίες και από αυτής της βάσης με τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων προετοιμάζουμε νέες κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή αυτών των εκθέσεων. Σε αυτή τη βάση τα δεδομένα θα ταιριάζουν σε μια νέα εκδοχή του συστήματος καταγραφής των παρατυπιών. Θέλω να σας ενημερώσω απλώς πως ε, αναμένουμε να είναι λειτουργικό το νέο αναβαθισμένο σύστημα το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Οι εθνικές στρατηγικές καταπολέμησης της απάτης τώρα. Όπως είπε ο εισηγητής, ε, φέρουμε υποχρεώσεις ε, όπως και τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν ένα και αποτελεσματικότερη δράση για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό φαίνεται από τον εντοπισμό αλλά και τη δίωξη περιπτώσεων 100 1649 υποθέσεις, ε, περισσότερες από το 2013 όμως θα πρέπει να βελτιώσουμε περαιτέρω αυτό το ποσοστό και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για τον εντοπισμό, την υποβολή αναφορών, τη δίωξη και την επιβολή κυρώσεων για τις περιπτώσεις απάτης, ούτως ώστε να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη αυτό που θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποτελεσματικές εθνικές στρατηγικές καταπολέμησης της διαφθοράς προς τα παρον είναι προαιρετικές. Πέντε κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει τέτοιες εθνικές στρατηγικές. Ενθαρρύνουμε και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Συνεργαζόμαστε δε με αυτά που έχουν ήδη υιοθετήσει τη στρατηγική τους ώστε να βελτιώσουμε και τη δράση που αναλαμβάνουμε στον τομέα της ανταλλαγής ε, βελτίστων πρακτικών ε, και εμπειριών. Ε, τρίτον, αφέρθηκε στις κρατικές προμήθειες ο Μετά την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τις κρατικές προμήθειες, η Επιτροπή επιδιώκει να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του, διαχειριστικού συστήματος για τις παρατυπίες δηλαδή και να υπάρχει υπάρχει διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων, ούτω ώστε να γίνεται βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών και φυσικά να ενισχύσουμε και τη διαφάνεια. Ξέρουμε ότι ο καλύτερο φίλο του φορολογουμένου είναι η διαφάνεια. Ό,τι περισσότερο πετύχουμε, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, δημοσιοποίηση των στοιχείων των δικαιούχων. Επίση, είναι σημαντικό, προβλέπεται εξάλλου από την νομοθεσία και τέτοιου είδου πληροφορίε θα πρέπει να δημοσιεύονται. Τέταρτο, των δείκτες για τη διαφθορά. Σε σχέση με τις στατιστικές και τους δείκτες διαφθοράς στα κράτη-μέλη υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τον ορισμό και την στατιστική καταγραφή των πρακτικών. Θα πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε και αυτό το ζήτημα μεσοπρόθεσμα ούτως ώστε να υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες για αυτό το ζήτημα και θα ήθελα να σας απαντήσω ναι ε, η διετής έκθεση κατά πολέμηση της διαφθοράς είναι κάτι που επίσης επεξεργαζόμαστε. Θα είναι έτοιμη το 2016. Πέμπτον, η που θα δοθεί σε συστάσεις σε εθνικό επίπεδο και η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Συμφωνούμε ότι η συνολική δίωξη των πατών και παρατυπιών κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ιδιαίτερη σημασία και στα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες ε, ούτως ώστε μεταξύ άλλων να υπάρχει υπάρχει και ενημέρωση για τις δράσεις που αναλαμβάνουν σε εθνικό επίπεδο. Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θεωρούμε ότι θα μας βοηθήσει. Σε αυτό το τομέα πιστεύουμε δε επίσης πως η αξιολόγηση ε, του κανονισμού 823 του 2003 σε σχέση με τις ε, έρευνες πρέπει να ολοκληρωθούν, έπρεπε να έχουν ολοκληρωθούν ε, και πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2017 θα μας βοηθήσει. Σε αυτό πιστεύουμε ότι η Ευρώπη το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα ο κανονισμός 823 θα, είναι εργαλεία που θα μας βοηθήσουν ε, να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Επίσης έχουμε την εντολή του ΕΦΚΟ, είναι ξεκάθαρη και πιστεύουμε ότι το ταχύτερο δυνατό θα πρέπει στα πλαίσια του Γκρέκου να προχωρήσουμε. Έχουμε το βέλτιστο δυνατό σύστημα, λοιπόν, μπορούσαμε να σχεδιάσουμε στη διάθεσή μα. Τέλο, στην Επιτροπή συζητήθηκε το τι μπορούμε να κάνουμε για την ε, ανεξαρτησία της ποπτική Επιτροπής ε, της Γραμματείας ε, στις 4 Μαρτίου στην Επιτροπή ελήφθη μία απόφαση και εγκρίθηκε μία πρόταση τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας της ΟΛΑΦ ούτως ώστε η γραμματεία ε, της Εποπτικής Επιτροπής ε, να μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί η πρόταση και από εσάς ε, το ταχύτερο δυνατό, ούτως ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε δυνατή σύγκρουση συμφερόντων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Λούνες που έχει το λόγο ε, για ένα λεπτό εκ μέρους Επιτροπής Εξωτερικού Μπορείου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αληθεύει όταν διασπαθίζονται χρήματα φορολογουμένων είναι πραγματικά έσχος ε, και όταν υπάρχουν και απάτες ε, και εδώ υπάρχουν αρκετές παρατηρήσεις σε αυτή την έκθεση. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Όλαφ ακόμα πιο έντονα να δράσουν. Όσον αφορά αυτά τα ποσά στην έκθεση, μας εκπλήσουν. Γνωρίζουμε όλη την ιστορία των ε, απατών όσον αφορά την πολιτική συνοχής ή όσον αφορά τις ενισχύσεις για τη γεωργία. Αυτή η έκθεση θα πρέπει σε προληπτικά μέτρα να επικεντρώνεται και να τα αναφέρει διότι στις απάτες είναι καλύτερο να προλαμβάνουμε τις απάτες παρά να θεραπεύουμε τον υστέρων. Τρίτον, η έκθεση τοποθετείται υπέρ ε, μιας νέας οργάνωσης, ευρωπαϊκής οργάνωσης. Ακόμα μια ευρωπαϊκή οργάνωση οργανισμός ε, παράλληλα με την Όλαφε. και διαρωτώ με, είναι πραγματικά αναγκαίος αυτός ο οργανισμός, δεν θα μπορούσαμε πιο αποτελεσματικά να δράσουμε. Δεν βλέπω τον επόμενο ομιλητή, ούτε τον κύριο Γέζεκ, ούτε τον κύριο Βόν. Οπότε θα πάμε στην κυρία Μπρεσό, εν ονόμα τη Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ κυρία Προέδρε. Προχωρούμε βιαστικά. Βλέποντας ότι λείπουν συνάδελφοι, θα ήθελα να επιθυμίσω ότι πρέπει να παραμείνει η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στα θεσμικά όρια τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και θα πρέπει να στερνιστούν το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους αυτό, το επίκεντρο της πολιτικής μας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Αυτό είναι κάτι που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαφθορά και η απάτη εις βάρος του προπολογισμού της Ενώσεω είναι, ε, είναι ευθέως ανάλογα με την διαφάνειας των μηχανισμών ανάθεσης και του τρόπου απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων. Θα πρέπει κατά την άποψή μου να γίνει σαφή διάκριση μεταξύ απάτης και σφαλμάτων και θα πρέπει να δίδονται πληροφορίες όσον αφορά τις απάτες αλλά και όσον αφορά τα συχνά σφάλματα παρουσιάζοντας και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα ούτω ώστε οι χρήστε των πόρων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως και οι αρχέ διαχείριση να είναι καλύτερα ενήμεροι και συνεπώς να είναι σε καλή τη θέση να διακρίνουν τη διασύνδεση μεταξύ απάτης και σφάλματος με τα αποτελέσματα. Ίσως και σφάλματα που οφείλονται σε κάποιες δυσκολίες και δυσκολίες που θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε. Να τις μειώσουμε με τη δραστηριότητα για την καλύτερη νομοθεσία. Με το μεταξύ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε να κάνουμε τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών ειδών προβλημάτων αυτό θα βοηθήσει πολύ τους χρήστες και θα μας επιτρέψει να βρούμε και ποιοι είναι οι πραγματικοί απαταιώνες σε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Μπαίνουμε στη συζήτηση. Εκ μέρους του ΕΛΚ η κυρία Πιτέρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σε σχέση με τα θεσμικά όργανα έχουν ως στόχο να διασφαλίζουν τα κονδύλια των φορολογουμένων. Είναι θεματοφύλακες για τη δαπάνη αυτών των κονδυλίων. Η καταπολέμηση οποιονδήποτε παρατυπιών θα πρέπει να είναι ανώτατη προτεραιότητα, διότι η διαφθορά και οι απάτες τροφοδοτούν και τις τρομοκρατικές οργανώσεις και το οργανωμένο έγκλημα και υπονομεύουν την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και της δημοκρατίας και έχουν επιπτώσει επιπλέον όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα την ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ωστόσο αυτή η μάχη είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Τα διοικητικά συστήματα διαφέρουν μεταξύ του. Θα έπρεπε να εργαστεί πραγματικά σκληρά με ένα συστηματικό τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάκτηση κονδυλίων και ποσών όσον αφορά του ίδιου πόρου και σε κοινού κανόνε και κανονισμού για τι αναφορέ Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και τα επιλεγμένα σχέδια θα πρέπει να οδηγούν στην ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει να προαχθούν επίσης κανόνες και κανονισμοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των πληροφοριοδοτών και να υπάρχει και πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Ωστόσο η πρόταση για την χρηματική υποστήριξη όσον αφορά τις, ε, τον διασυνοριακό, ε, τις ε, διασυνοριακές δημοσιογραφικές δραστηριότητες ε, θα αποδυναμωνόντουσαν αν δεν ε, διετίθεντο κονδύλια. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί. Κύριος Πυρίνσκι, για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες για ένα δίλεπτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Χρησιμότατη διαδικασία καταρτήσεως εκθέσεως και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι τέτοια που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση εμπιστοσύνης των πολιτών. Δηλαδή να πιστεύουν ότι προστατεύονται σωστά τα οικονομικά του συμφέροντα. Θέλω να αναφερθώ σε τρία σημεία που περιέχονται στην έκθεση και να ζητήσω από τον Επίτροπο να σχολιάσει. Πρώτα απ' όλα, οι διακοπές και οι αναστολές. Είναι σημαντικό να τονίσουμε τι εμπεριέχεται στην έκθεση ότι αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την σχετική νομική βάση και στο πλαίσιο, κυρία Αντιπρόεδρε, ενός σημαντικοτάτου στοιχείου. Έχετε υιοθετήσει ένα νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και θα ήθελα να σας καλέσω να μας πείτε ποια είναι η προσδοχία σας για ένα ολιστικό σύστημα έγκυρης ε, έγκαιρο εντοπισμού και ε, αποκλεισμού που θέλει να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι η πρόληψη, η πρόληψη είναι το σημαντικό στοιχείο. Δεύτερον, τον άμεσα, το θέμα της άμεσης διαχείρισης των πόρων, κύριε Επίτροπε, είναι ανησυχητικό, διότι έχουμε μεγάλη αύξηση των απατών και των ατασταλιών το 2014. Θέλουμε λεπτομερείς εξηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Και να μας πει τι δράση σκοπεύει να αναλάβει. Τρίτον, αναφερθήκατε στη σωστή ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων. Συμφωνώ με τους συναδέλφους και με το περιεχόμενο της εκθέσεως. Η κατάσταση είναι άκρο ανικανοποιητική. Δεν έχουμε αρκετά σαφή εικόνα. Βασιζόμαστε πολύ στις προσπάθειες που αναφέρατε, ούτω ώστε να κάνουμε αλλαγές και για την έκθεση του επόμενου έτους ακόμα. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ η κυρία Μακοβέη για το ECR, για ένα δίλεπτο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Το 2014 τα κράτη-μέλη ανέφεραν πάνω από 1.600 περιπτώσεις απατών περίπου 540 εκατομμυρίων ευρώ έγινε λόγος για τέτοιου είδους ε, παρατυπίες. Ε, δεν είναι λεπτομέρειες και παρονυχίδες, είναι χρήματα των φορολογουμένων, δικά μας χρήματα. Πρέπει να υπομειστεί πλήρως ε, τις ευθύνες της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάκτηση αυτών των ποσών. Επίσης πρέπει να εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες για την ανάκτηση πληρωμών ή την διακοπή κιόλα πληρωμών. Για την περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Είναι ένα από τα κατεπήγοντα μέτρα, ελάχιστα μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν και να δράσουμε από ένα άλλο μέτρο είναι η προστασία των πληροφοριοδοτών. Η πείρα τη διδάσκει είδαμε ότι όσοι εργάστηκαν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και είναι πληροφοριοδότες, εκείνοι οι οποίοι δηλαδή στιγμάτισαν τις περιπτώσεις ε, των ε, καταχρήσεων βρίσκονται σε δινή κατάσταση και όταν χάνει χρήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προστατεύονται αυτοί οι άνθρωποι ώστε να μπορούν να προστατευθούν τα κονδύλια. Ε, μετά έχουμε και τις συμφωνίες με τις καπνικές εταιρείες. Όλες αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να, είναι δημο, να δημοσιευθούν, να δημοσιοποιηθούν στο μέτρο του δυνατού, στο ευρύτερο δυνατό μέτρο, ώστε να καταφέρουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να αντιμετωπίσουμε το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού αποτελεσματικά. Επίσης ε, η οδηγία θα πρέπει να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε όλων των ειδών της ε, παρατυπίες. Η, τα κράτη-μέλη σε σχέση με τον ΦΠΑ, το ΦΠΑ που πρέπει να μπορέσουν να πιστούν να αντιμετωπιστεί ως ε, περίπτωση αδικήματος ή ως έγκλημα. Επίσης Επίσης ε, η ρύθμιση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλα τα χρήματα θα πρέπει να καταλήγουν, να δούμε ότι καταλήγουν σε ένα κορβανά. Αν κλέβονται από ένα κράτος μέλος είναι εις βάρος όλων μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλή, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Γεωργίευα, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον εισηγητή Γιαβόρ για την εξαιρετική έκθεση και ευχαριστώ και την Επίτροπο Γεωργίευα για την ε, διεξοδική εναρκτήρια παρουσίαση που έκανε. Ε, πλήττεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις παρατυπίες. Ε, χρειαζόμαστε μέτρα για να προστατεύσουμε το της ευρωπαϊκή Η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων ε, απηχεί όλα τα διορθωτικά μέτρα ε, που χρησιμοποιούνται ούτω ώστε να προστατευτεί ο προϋπολογισμός από παρατυπίες, απαράτυπες επληρωμές και ατασταλίες. Τα... Είναι κοινή αρμοδιότητα των κρατών μελών η προστασία των οικονομικών συμφερόντων και η καταπολέμηση της απάτης είναι ζωτική σημασία συνεργασία των κρατών μελών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Η Επιτροπή εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση όπως ακούσαμε και από την Αντιπρόεδρο Γεωργίευα. Βλέπουμε την κατάσταση στον τομέα των οικονομικών συμφερόντων μέσα στην έκθεση για τον εντοπισμό, την υποβολή αναφορών ε, για τις παρατυπίες, ε, για ε, τις δαπάνες και τα έσοδα. Επίσης εντοπίζονται και παρασιάζονται διάφορα μέτρα ως προς τη διεξαγωγή ελέγχων. Ένα κοινό σύστημα επίσης δικτώνει για να μετρηθεί το επίπεδο διαφθοράς στα κράτη-μέλη, τροποποίηση του κανονισμού για την προστασία των whistleblowers και στον τομέα των ε, κρατικών ε, ε, προμηθειών κατά πολέμηση του λαθρεμπορίου και της παραποίησης προϊόντων Οποιαδήποτε δόλια δράση βάρος των οικονομικών συμφερόντων ε, αναφέρεται μέσα στην έκθεση και ε, ε, αναφέρεται ότι πρέπει να λειτουργούμε βάσει αρχής αποτελεσματικότητας των μέτρων που αναλαμβάνουμε. Φυσικά θα πρέπει να μην αποθαρρύνουμε τους δικαιούχους κατά το σχεδιασμό των νέων μέτρων. Η Πρόεδρος διακόπτει τον κύριο Αλή, θα συνεχίζει ο κύριος Αλή, θα πρέπει να συνεχίσουμε τους ελέγχους προστατεύοντας τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον θεσμό της. Ευχαριστούμε κύριο Σβαλή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν οι κυβέρνηση που λέγονται ότι είναι φιλοπροπιστικές πρέπει να θετούν μέτρα για την προστασία των φορολογωμένων των Ευρωπαίων ε, γίνονται αμέσω σκεπτικιστές γι' αυτό. Η δαπάνη των χρημάτων στη σκιά οδηγεί στο να λαμβάνονται σημαντικέ αποφάσει για τα αλλαγή πληροφοριών, συνεργασία και διαφάνεια που περιέχονται στην οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε πλέον να παραθέτουμε εύκολε δαπάνε και απάτε και να τα δεχτούμε. Τι δαπάνε. Η έλλειψη διαφάνεια όσον αφορά την τεκμηρίωση, όσον αφορά του διαγωνισμού που ανατίθενται άμεσα τα έργα. Οι εθνικοί έλεγχοι δεν διεξάγονται σωστά και υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και κυρίω υπάρχει ελάχιστη βούληση των κυβερνήσεων να συνεργαστούν σε θέματα ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα φορολογικά και τα τραπεζικά δεδομένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αποτελεθεί πραγματικά η μεγάλη φοροδιφυγή και η φοροαποφυγή και η ανακύκλωση του χρήματο. Βλέπουμε ότι το Λουξεμβούργο του Ιούνκερ ότι ήταν πρωταθλητή σε αυτό το θέμα. Ε, και είναι σκανδαλώδη η έλλειψη διαφάνεια όσον αφορά και το πρόγραμμα για τη σύνδεση Τωρίνου Λιών. Λοιπόν, και δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα όσον αφορά τα έργα που χρησιμοποιούνται από ευρωπαϊκού πόρου και θέλουμε που παίρνουν αρνητικέ αποφάσει. Πρέπει να δώσει λύση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Βάλη. Ο κύριο Συναδεινό, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, είναι σημαντικό να θεσμοθετούμε την ύπαρξη και λειτουργία υπηρεσιών και μηχανισμών για την καταπολέμηση τη απάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικότερο όμω είναι να λαμβάνουμε υπόψη τα αποτελέσματα των εκθέσεων και των συμπερασμάτων για τη χάραξη πολιτικών και του τρόπου αντιμετώπιση των κακών κειμένων για παράδειγμα είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη η απλούστευση των κανόνων και διαδικασιών που αφορούν τι δημόσιες δαπάνες και τα έσοδα από ίδιους πόρου ώστε να περιοριστούν οι μη δόλιε παρατυπίες που για το 2014 ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 362 και 176,2 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Όμως αυτονόητη και επιβεβλημένη είναι η αναθεώρηση τη απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την παροχή βοήθεια ύψους 3 δι ευρώ στην Τουρκία όταν η έκθεση για την καταπολέμηση της απάτης επισημαίνει ότι αυτή αποτελεί το βασικό πρωταγωνιστή των εξόφθαλων παρατυπιών που συνδέονται με τα κονδύλια προενταξιακής βοήθειας και κυρίως εκείνα που σχετίζονται με τη διασυνοριακή συνεργασία. η ένωση κινείται στα όρια της δολιότητος όταν η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά στην αξιοπιστία της τουρκίας. οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ηγέτες των κρατών μελών ακόμη πιστεύουν ότι δίνοντα κονδύλια θα περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές στην ευρώπη. πόσοι ακόμη θέλετε να σας πούν ότι η τουρκία είναι απατεώνας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μιλούσατε πάρα πολύ γρήγορα και άργησε η μετάφραση. ένα 1,5 ε, λεπτό παρακαλώ. Αξιότιμη Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Γεωργίευα, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Γιαβόρ, τον εισηγητή, για την διεξοδικότατη έκθεση που συνέταξε. 150 δις χρήματα φορολογουμένων. Αυτός είναι περίπου ο προϋπολογισμός της Ένωσης. Δικαίως θέλουν οι φορολογούμενοι να ε, γνωρίζουν ότι δεν ε, διαπράττονται απάτες ε, με αυτά τα χρήματα. Το 2014 ε, 538 εκατομμύρια των εσόδων σχετίζονται με περιπτώσεις απάτης. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να φέρουμε διορθώσεις. Έλεγχος των δαπανών και ε, ε, επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση απάτης. Για να γίνει αυτό Τρία είναι τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λειτουργεί προορατικά και να παρακολουθεί την εκταμίευση και τη χρήση των κονδυλίων. Ως εκ τούτου, δεύτερον, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λογοδοτούν ε, σε σχέ... μετά την παρακολούθηση των προγραμμάτων και την παροχή σωστών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτον θα πρέπει για την καταβολή τη απάντηση να έχουν ένα κοινό στόχο τα κράτη-μέλη. Τελικά ε, έτσι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτόν τον στόχο που επιδόκουμε εδώ και χρόνια, δηλαδή τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, ΕΠΟ. Ελπίζω να μας ακούνε τα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούει αυτά που τις λέμε. Ευχαριστούμε κύριε Σάρβαμα. Έχετε μια γαλάζια κάρτα. Τη δέχεστε ο κύριος Σορβίτς. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον συνάδελφο Σαββάμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την Όλαφ τι πάει στραβά και η Όλαφ δεν μπορεί να έχει τις επιδόσεις που χρειάζονται. Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο οργανισμό εδώ ή μήπως θα πρέπει να ξανασχεδιαστεί εξ αρχής η Όλαφ. Δεν ναι. ε, υπήρξε η μετάφραση, αλλά μάλλον και εσείς καταλάβατε, Πρόεδρε, ότι ρώτησε ο κύριος Ρίμπη γιατί χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό εισαγγελέα. Συγχαρητήρια στο γερμανό μου δάσκαλο. Μα, ε, υπάρχει αρμοδιότητα, δικαιοδοσία ε, στα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση της απάτης ε, και οι εθνικές αρχές ξέρουν ότι δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα σύνορα. Υπάρχει ένα κενό ε, στις περιπτώσεις διασυνοριακής απάτης και περιμένουμε 15 χρόνια να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ελπίζω τώρα να γίνει. Ευχαριστούμε. Αγέλα Σέντερ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, έχουμε για άλλη μια φορά εφέτος αυτή τη συζήτηση για ένα προϋπολογισμό που είναι όλο και πιο πενιχρός και επισφαλής και με όλο περισσότερες πιέσεις, περισσότερες φιλοδοξίες. Γι' αυτό ευχαριστώ τον κύριο Γιάβορ που έκανε, υπογράμμισε ιδιαίτερα την προστασία των εσόδων που είναι σημαντική υπόθεση και που εφέτος δεδομένης της ε, απάτης ε, σε σχέση με το ΦΠΑ σε σχέση με το 2013 ήταν 188 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περισσότερο από τον προϋπολογισμό του 2016 και αυτό είναι κάτι το ανέφικτο το να διατηρηθεί και πρέπει να εστιαστούμε σε αυτό μέσω της Όλαφ αλλά και της οδηγίας ΠΙΦ να συμπεριληφθεί το ΦΠΑ ως περίπτωση κατεπηγόντως ε, όσο το δυνατόν γοργότερα. Υπάρχει κατεπήγον να καταπολεμήσουμε αυτές τις απάτες που είναι πάρα πολύ μεγάλα ποσά για ένα προϋπολογισμό που είναι πενιχρός. Και το ίδιο διακόπτεται. Δεν είχα δύο λεπτά. Μόνο ένα, εντάξει, ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη. Κρίμα, ο κύριος Άρνοτ. Ένα Εάν μιλάμε για την καταβολέμηση της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε χάνουμε δισεκατομμύρια σε παρατυπίες φεύγουν και από τον εντοπισμό μέχρι την ε, υποβολή αναφορών περνάνε τρία χρόνια και τέσσερις μήνες. Ε, ε, έχουμε ίδιους σπόρους Ε, και μιλάμε για την απάτη του ΦΠΑ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι είναι ένα και πιο γραφειοκρατικό το σύστημα για την ε, συλλογή των φόρων. Δεν υπάρχει προηγούμενο είναι ανήκωστο το πόσο γραφειοκρατικό είναι και τώρα ζητάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί και στην επινική δικαιοσύνη να υπάρξει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μα τι παράδειγμα θα δώσουμε υποτίθεται. Ε, κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα θέλουμε όλο ένα και περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση για να το λύσουμε. Εάν ήξεραν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι άνθρωποι τι γίνεται εδώ πέρα και το τι ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, ψήφιζαν ε, στο δημοψήφισμα ψηφίσμα για να βγει οριστικά το Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε ο κύριος Δεντόφσκι. Ε, μισή λεπτό λέει γαλλιστή. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Επίτρεπε. Είναι σημαντικό να δράσουμε ενεργά, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για αυτά που συζητούμε. Αλλά σε σχέση με τη δική μας άποψη από πλευρά του ΕΛΚ πρέπει να πω ότι είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Η διαφθορά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και έχει επιπτώσεις ε, στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι εις βάρος των συμφερόντων των πολιτών μας. 120 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτά τα οποία χάνουμε. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα η καταπολέμηση αυτής της διαφθοράς. Όμως ε, είναι ένα θέμα που αφορά όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και κάθε κράτος μέλος και θέλω να το τονίσω αυτό. Πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά είναι η παριθμόν ένα μάστιγα και πρέπει να καταπολεμηθεί με κάθε τρόπο, με αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δίνουν ε, την δυνατότητα να, να δαπανούν τα κονδύλια αυτά με τον πιο υπεύθυνο τρόπο και να υπάρχει διασφάλιση ότι η μέγιστη αξία, πρόσθετη αξία θα επιτυγχάνεται από την χρήση αυτών των κονδυλίων. Αν δεν χρησιμοποιούμε λοιπόν αποτελεσματικά τα κονδύλια θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Είναι ένα πολύ ισορροπημένο κείμενο το κείμενο της έκθεσης, ε, ποιοτικά αναβαθμισμένο και θέλω πραγματικά να τονίσω όλοι θα πρέπει να εμπλακούν με τον πιο ενεργό τρόπο και να δράσουν ώστε να εφαρμοστούν οι προτάσεις αυτές. Σας ευχαριστώ και εγώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Νομίζω ένα σημαντικό ζήτημα είναι το ότι βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη, αναγκαιότητα να προστατεύσουμε τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όχι μόνο προφανής αυτός ο στόχος, αλλά είναι σημαντικό να καταδείξουμε ότι τα κονδύλια των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά είναι κοινό ο στόχο, κοινό το συμφέρον να προστατευτούν τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προστασία αυτή για να επιτευχθεί πρέπει όλοι να υπομισθούμε τι ευθύνε μα στη δράση μα, Ξεκινώντας, με την σωστή και πιο ορθολογική δαπάνη των διαθέσιμων κονδυλίων. Αν συνεχίσουμε να, να αντιμετωπίζουμε το θέμα των δαπανών ε, σαν κάτι επουσιώδες, ε, δεν θα λειτουργήσει με κανένα τρόπο το σύστημα πρέπει να δούμε ότι πάνω από 100 εκατομμύρια με, παράτυπο τρόπο χρησιμοποιήθηκαν. Винаги съм Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην αντικειμενικότητα, στο σκοπό δηλαδή να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα των πολιτών. Στην έκθεση όμως ότι βλέπουμε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον που διαπιστώνεται. Βλέπουμε ότι χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση, η οποία κοινή προσέγγιση περνά μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χαιρόμαστε που βλέπουμε τη διαφορά που γίνεται μεταξύ απάτης και σφάλματος. Τα σφάλματα οφείλονται στις επαχθείς διαδικασίες και πολύ συχνά οι δικαιούχοι προτιμούν να πάρουν μια εθνική πίστοση παρά να απευθυνθούν προς τα ευρωπαϊκά ταμεία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε σαφέστερους και απλούστερους κανόνες. Χαίρομαι που βλέπω ότι η χώρα μου αναφέρθηκε ως μια χώρα η οποία παρουσίασε με σωστό τρόπο τα σφάλματα, ακόμα και πριν τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι που βλέπω επίσης και το έργο που κάνει η Επίτροπο στον τομέα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρία Γεωργίευα, η έκθεση αυτή ήμουνα για την έκθεση του 2013 εισηγητής και βλέπω ότι δεν μειώθηκαν οι περιπτώσεις απατών αλλά αυξήθηκαν και για το 2014 χάσαμε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ ε, όμως μόνο μικρό ποσοστό αυτού του ποσού ανακτάται από τα κράτη-μέλη. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι τα κράτη-μέλη παραλαμβάνουν πολλούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν υπέχουν υποχρέωση να παράσχουν ε, σωστά στοιχεία, καλά στοιχεία όσον αφορά την χρήση των πόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπώς πρέπει να ετοιμάσει ένα καλό σύστημα για την παροχή πληροφοριών, οι οποίες πληροφορίες θα μας επιτρέπουν να δούμε πώς εφαρμόζουν τις συστάσεις όλα αυτά κάτι μέλη και πώς χρησιμοποιούν τους πόρους. Η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο στην ανάκτηση των χρημάτων. Πάμε τώρα στην προσέλκυση της προσοχής του, της Προέδρου με τον κύριο Πόσπισιλ. δικασία κάτσε με άλλα λόγια. Κύριε Πόσπισιλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ προσεκτικά άκουσα τις παρατηρήσεις της κυρίας Επιτρόπου Γεωργίευα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην καταπολέμηση των παρατυπιών και όσων έχουν και τεχνικό χαρακτήρα και παρατυπιών που εκ παραδρομής ε, σημειώθηκαν. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό από πλευρά της, ε, του οργανισμού για την ε, εισαγγελία. Εργάστηκα σχετικά με την Σεχία για αυτό το θέμα και πάντα είναι κάτι το οποίο συναντούσε και αντίσταση. Ας μην αυταπατώμεθα θεωρώντας ότι αυτός ο νέος οργανισμός ε, θα επιλύσει το πρόβλημα αυτομάτως. Κάνουμε λόγο για παρατυπίες ε, και πρέπει να δούμε ότι υπεύθυνα θα πρέπει να είναι τα εθνικά δικαστήρια. Ακόμα και αν ενεργοποιηθεί η εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα πρέπει τα εθνικά δικαστήρια τα οποία θα είναι υπεύθυνα να δράσουν ώστε σε συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών να καταπολεμηθούν αυτές οι περιπτώσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι είναι σημαντικότατη η έκθεση. Λαμβάνει υπόψη το επίπεδο των απατών στα κάτι μέλη. Η απάτη οδηγεί σε διαφθορά και η διαφθορά επηρεάζει τους πολίτες των κρατών μελών. Δημιουργεί κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Η διαφθορά μπορεί να συμβάλλει στη χρηματοδότηση των ε, δραστηριοτήτων τρομοκρατικών δικτύων και η διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία. Πρέπει να βελτιώσουμε τους ελέγχους, αλλά και η πρόληψη είναι ακόμα πιο σημαντική θα έλεγα. Είναι πρόβλημα για τους πολίτες μιας χώρας όταν υπάρχει περικοπή των ε, πληρωμών ή αναστολή των πληρωμών λόγω σφάλματος που διαπιστώνεται. Ε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε απλουστευμένες διαδικασίες διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά σφάλματα ε, όσον αφορά τις δαπάνες και όσον αφορά και την ε, αναφορά των προβλημάτων. Δεν πιστεύω στη δημιουργία νέων θεσμών. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε την πρόληψη. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Σύμφωνα με την έκθεση, ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διασφαλιστεί μέσω τη Όλαφ, η οποία έχει σαν ρόλο να εντοπίζει και να διερευνά περιπτώσει απάτη και διαφθορά, καθώ και άλλε παράνομε δραστηριότητε ωστόσο το σύνολο των παρατυπιών που αναφέρθηκαν για το 2014 ανέρχεται περίπου σε 3,24 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ ο δημοσιονομικό αντίκτυπος των παρατυπιών που δηλώθηκαν είναι κατά 36% μεγαλύτερο μεγαλύτερος σε σχέση με το. 2013. επιπλέον η Όλαφ, ενώ έχει συσταθεί από την ευρωπαϊκή ένωση προκειμένου να πατάξει τη διαφθορά και την απάτη εντός των κρατών μελών τη, δεν κάνει τίποτε για να συμβάλλει επιβοηθητικά στην πάταξη της φορολογικής απάτης που λαμβάνει η χώρα στην ευρωπαϊκή ένωση καθώς και στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής των πολυεθνικών εταιριών σε φορολογικούς παραδείσους και τη μεταφορά κερδών τους σε αυτές. είναι επομένως αναγκαίο η όλαφ να συμβάλλει πιο ενεργά κατά της φοροδιαφυγής των πολυεθνικών και να συμβάλλει έμπρακτα στην καταπολέμηση κάθε παράνομης δραστηριότητας που πλήττει την ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σόλτε, ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Γιάβορ για την πολύ καλή συνεργασία σε σχέση με αυτή την έκθεση. Δύο προβλήματα θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, το αθέμητο εμπόριο. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα βέβαια και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χάνουν πάρα πολλά έσοδα από πλευρά τους λόγω του αθέμητου εμπορίου. Μέχρι 37 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις και πρέπει φυσικά για τους Ευρωπαίους φορολογουμένους να δράσουμε αποτελεσματικά. Έχουμε μετά και το θέμα των δημόσιων πληρωμών και των παραγγελιών. Και εδώ διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σφάλματα και παρατυπίες. Και φυσικά μπορούμε να υπολογίσουμε ποιο είναι το ύψος, πώς δηλαδή με αυτά τα ποσά ε, βλάπτεται, υπονομεύεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και πρέπει να αναλυθούν μέτρα κατά αυτής της κατάστασης. Όμως το όνειρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πόρο απέχει ακόμα από την πραγματικότητα. Τα αρμόδια κράτη-μέλη πρέπει να πράξουν περισσότερα πρώτα. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είπατε, Επίτροπε, ότι η διαφάνεια είναι ο καλύτερος φίλος του φορολογουμένου. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι και ο καλύτερος φίλος της καταπολέμησης της διαφθοράς και γι' αυτό είναι σημαντικό ε, τον 21ο αιώνα να μεριμνούμε ώστε όλα τα κράτη-μέλη με ένα κλικ ε, στο διαδίκτυο να γνωρίζουν ακριβώς ε, ποιος ήταν ο αποδέκτης κάθε πληρωμής, ε, ποιος είναι ο κάθε δικαιούχος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε την απάτη, να αποτρέψουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων και την κατασπατάλη στη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να υπάρξει εκπαίδευση και να έχουμε μια βάση δεδομένων για τους δικαιούχους της πολιτικής συνοχής για να εντοπίζουμε ευκολότερα ε, και να αποτρέπουμε τις παρατυπίες. Ε, σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνεται με την κυρία Μάλετιτς η διαδικασία ε, Catch the Eye. Θα επιστρέψουμε τώρα στην Αντιπρόεδρο Γεωργίευα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα σχόλια και τις συστάσεις που κάνατε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα κυρίως που υποβάλλατε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, πρόληψη. Όπως είπε ο κύριος Πυρίνσκι, Τώρα θεσπίζουμε συστήματα, μηχανισμούς έγκυρης προειδοποίησης, χάρη στα οποία μπορούμε να ενοποιούμε τα στοιχεία από διάφορες βάσεις δεδομένων, το ακούσαμε και στην προηγούμενη, σε αυτή την τελευταία παρέμβαση, για να ξέρουμε από πού προέρχονται τα χρήματα, ποιος είναι ο δικαιούχος και να ε, έχουμε ολόκληρη ε, την πορεία της πληρωμή. Ε, δεν επικοινωνούν όλες οι βάσεις δεδομένων αυτή τη στιγμή και γι' αυτό εστιάζουμε την προσοχή μας στη ρύθμιση αυτού του προβλήματος. Στην πρωτοβουλία για την επίτευξη αυτών αποτελεσμάτων επιδιώκουμε ένα τρόπο να βλέπουμε όχι μόνο την πορεία των χρημάτων αλλά και το αποτέλεσμα, το, το τι αποκομίζουμε ε, από την πληρωμή αυτή. Θα χρειαστεί χρόνος και χρειάζεται ενοποίηση των επιμέρους προσπαθειών, αλλά όπως σας είπα, ήδη ε, το επόμενο τρίμηνο θα υπάρξει καλύτερη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων. Δεύτερον, ακούστηκε πόσο σημαντικό είναι να διαχωριστούν οι απάτες από τις παρατυπίες. Φυσικά, η απάτη είναι ένα καρκίνωμα της κοινωνίας ε, από τα πιο επικίνδυνα. Είναι όμως δύσκολο και να εντοπιστεί διότι σε κάθε δόλια δραστηριότητα ε, πολύ φαιά ουσία και χρήματα ε, στοχεύουν στην απόκρυψη της δραστηριότητας. Τι μπορούμε να κάνουμε. Απλούστευση των κανόνων ώστε να είναι δυσχερέστερο να υπάρξει παραπληροφόρηση και απόκρυψη. Έτσι, σίγουρα θα περιορίσουμε όχι μόνο την απάτη, αλλά και τις παρατυπίες. Δεύτερον, στην ανάλυση που κάνουμε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι γίνεται μετά τον εντοπισμό της απάτης. Ε, δηλαδή, πέρα από τον εντοπισμό της, ε, πώς ε, θα, πώς ε, θα προλαμβάνουμε τις ε, απάτες και τις παρατυπίες. Τρίτον, σε θεσμικό επίπεδο, ενώ ξέρουμε από τη δουλειά της Όλεφ ότι υπάρχουν παρατυπίες και δόλιες παρατυπίες, απάτες, μας λείπει το σφυρί, δηλαδή στέλνουμε εμείς τις προφορίες στα κράτη-μέλη και πρέπει στη συνέχεια να κινηθούν τα κράτη-μέλη. Εκεί που είναι ισχυρό το νομικό σύστημα τότε αναλαμβάνεται δράση, εκεί όμως που υπάρχουν κολλήματα νομικά ενδέχεται και να μην αναλυφθεί η δράση. Κάποιοι αναφέρθηκαν σε αυτά μόνο 24 τις 100 και εδώ μιλάμε μόνο για δόλες αλλά και μη δόλες παρατυπίες διώκονται τελικά. Ε, γι' αυτό και σας μίλησα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα έχουμε το ε, σφυρί, ε, την δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. Έχει αποδυναμωθεί η αρχική πρόταση, ομολογουμένως έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας. Η απάτη ΦΠΑ φαίνεται ότι έχει αποκλειστεί πλέον από την εντολή του ε, Ευρωπαϊκού Εισαγγελέου και φυσικά ένα μεγάλο κομμάτι ε, η ονία πάτης αποκλείεται από τη δράση του κατά αυτόν τον τρόπο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει με σαφήνεια να διαπραγματευτούν για την ε, εισαγγελία και θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα πρέπει να είναι μια προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι αυτός σκοπός οι θεσμοί. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικότεροι στην δράση μας. Αυτό επιδιώκουμε. Επίσης, κάτι σημαντικό που ακούστηκε είναι ότι είναι σημαντικό να ακούγονται οι φωνές των καταγγελόντων. Αυτό το κάνουμε για το προσωπικό μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το τι μπορούμε να κάνουμε είναι το ερώτημα για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τη δική τους εθνική νομοθεσία για τους καταγγέλοντες ποια είναι η δική μας ευθύνη. Θέλουμε να είμαστε συνετοί, δεν θέλουμε να υπερβούμε το πεδίο αρμοδιοτήτων μας. Ακούσαμε και το σχετικό σχόλιο ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η εθνική κυριαρχία και η επικουρικότητα. Ουδάλλως ε, μπορεί να, η ζημιά να ε, υπερσκελίσει το όφελος και φυσικά θα πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτού. Θα ήθελα, κύριε Πυρίνσκι, του χρόνου να έχουμε μια πολύ καλή ανάλυση σχέση με την αύξηση του ποσοστού των δολίων ε, παρατυπιών. Εντοπίζουμε περισσότερες ε, απάτες ή υπάρχουν περισσότερες απάτες. Αυτό θα πρέπει να διαπιστώσουμε και έχουν ήδη δρομολογηθεί σχετικές δράσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Ο συγητής, ο κύριος Γιαβόρα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για όσα είπατε και για την ε, πολύ αποδοτική συζήτηση την αποψηνή Εν συντομία, να πω εν είδη αντιδράσεως τα υποθέντα, πιστεύω ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτο στοιχείο, που συνδέεται και με την πρόληψη. Είναι η πλήρης διαφάνεια. Δεν υπάρχει απάτη, δεν υπάρχει διαφθορά όταν υπάρχει διαφάνεια. Αυτό αφορά και το μητρό για τις ομάδες πίεσης, το υποχρεωτικό μητρό για την καταχώρηση των, λομ, αλλά υπάρχουν και άλλες στοιχείες που αφορούν τη διαφάνεια. Χρειάζεται και καλύτερη υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων από τις εθνικές αρχές. Δεύτερον, χρειαζόμαστε αυξημένη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Η κυρία Μακοβέη το ανέφερε ότι η απάτη δεν καταπολεμάται χωρίς καλή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και των αρχών αυτών. Κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Τρίτο στοιχείο. Χρειαζόμαστε ισχυρούς θεσμούς. Όταν αφαιρόμαστε στην Όλαφ Μπορούμε να επικρίνουμε την Όλαφ βεβαίως, αλλά η Όλαφ δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς ε, τα δικαιώματα που απαιτούνται, τη δικαιοδοσία που πρέπει να έχει για να είναι ισχυρή. Πρέπει να ενισχύσουμε την Όλαφ. Να, ελέγχει το πώς, να ελέγχουμε πώς υλοποιούνται οι συστάσεις της Όλαφ τα κράτη-μέλη. Και χρειαζόμαστε και άλλους θεσμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Και μετά τελευταίο θέμα είναι οι κυρώσει. Εδώ υπάρχουν σοβαρά κενά από πλευρά ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πώς μπορούμε να υποχρώσουμε τα κράτη-μέλη να σέβονται τους κανόνες μέσω κυρώσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την διαφθορά και την απάτη. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Έχουμε προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς μια κμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα.